Ασπίζονται. Εμείς όμως δεν το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν για να έχουμε και μια καλή συμφωνία με την Ρωσία. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και για την επικοδομητική συνεργασία πρόεδρος. Σε ευχαριστούμε Χάνες. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου αυτή έκθεση και τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ολοκληρώνεται λοιπόν τώρα με αυτή την παρέμβαση αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η ψήφιση θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΥΠΑ της Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Με πληροφορούν ότι ο ρόλος, η θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου θα εκπροσωπηθεί σε αυτή την περίπτωση από την αγαπητή συνάδελφο κυρία Ερατό Ζάκου Μαρκούλη, ε, Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την καλωσορίζουμε, είναι αυτονόητο, στην Ολομέλειά μας, στην αίθουσα της Ολομέλειας. Για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση έχετε τον λόγο κυρία Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για να μας παρουσιάσετε την δήλωση αυτή. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Honorable Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, όλοι παρακολουθούμε με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία την ε, ε, εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε βίε συγκρούσει κατά τη διάρκεια ε, διαδηλώσεων που είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετού θανάτου και πολλού τραυματισμένου. Η κατάσταση ανάμεσα στου υποστηριχτέ του Πρόεδρου Μόρση και τη αντιπολίτευση του Εθνικού Μετώπου Σωτηρίας ε, φαίνεται ότι έχει ε, πλοκαριστεί ε, και, και τα δύο στρατόπεδα καλούν σε νέες διαδηλώσεις. Ζητώ συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Μία αγωνιώδης ερώτηση που έρχεται στο μυαλό είναι τι ε, γίνεται με την δημοκρατική μετάβαση της Αιγύπτου. Τη Δευτέρα συζητήσαμε την κατάσταση στην Αίγυπτο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνει αποκλιμάκωση της κατάστασης και ένας διάλογος χωρίς αποκλεισμούς για να βρεθεί μια λύση που να βασίζεται στην ε, συνένεση και που να αισθάνονται όλοι ότι εκπροσωπούνται. Προφανώς η Αίγυπτος χρειάζεται ένα ισχυρό σύνταγμα το οποίο να ε, αντιπροσωπεύει όλους τους Αιγυπτίους. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να ανακεφαλαιώσω κάποια από τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την τόσο διχαστική πολιτική κρίση. Στις 22 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Μόρση ε, εξέδωσε μια συνταγματική διακήρυξη όπου μεταξύ άλλων πραγμάτων έθετε την Προεδρία του υπεράνω του δικαστικού ελέγχου. Στις 30 Νοεμβρίου υιοθετήθηκε ένα σχέδιο συντάγματος από την ε, συντακτική συνέλευση όπου κυριαρχούν οι Ισλαμιστές και παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο και ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ένα δημοψήφισμα για το Σύνταγμα αυτό στις 15 Δεκεμβρίου. Ακολούθησαν ε, διαδηλώσεις και από τα δύο στρατόπεδα, αρχικά ειρηνικές, αλλά κατά λυπηρό τρόπο ε, οδήγησαν σε βίες εκδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος Μόρση απευθύνθηκε στο έθνος και ζήτησε διαπραγματα... Ε, συνομιλίες. δεν μετακινήθηκε όμως από την συνταγματική του διακήρυξη και κράτησε και την ημερομηνία του δημοψηφίσματος το Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας, δηλαδή το βασικό μπλοκ της αντιπολίτευσης που αποτελείται από φιλελεύθερα και λαϊκά κόμματα μεταξύ των οποίων ε, δεν υπάρχουν και οι υποψήφοι για πρόεδροι Άμρου Μούσα και Μοχάμεντα Ε, το Εθνικό λοιπόν Μέτωπο Σωτηρίας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες, ε, μια που κανένα από τα αιτήματά του δεν, ε, είχαν, ε, δεν είχε ικανοποιηθεί. Δηλαδή, απόσυρση της δήλωσης αυτής, ακύρωση του συνταγματικού δημοψηφίσματος και δημιουργία νέας συντακτικής συνέλευσης. Το Σάββατο έγινε ένας διάλογος με τη συμμετοχή 60 πολιτικών προσωπικότητων, χωρίς όμως τη συμμετοχή του Εθνικού ε, Μετώπου Σωτηρίας. Ο πρώτος Μόρση, μετά από τις συνομιλίες αυτές, ε, ακύρωσε την αρχική συνταγματική του διακήρυξη, ε, αλλά κράτησε την ημερομηνία για το δημοσίσμα την ίδια ε, νέες ε, διαδηλώσεις ακολούθησαν και των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Μόρση, αλλά η κατάσταση είναι πιο ήρεμη στους δρόμους. Το Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συμμετάσχει ε, στο ε, δημοψήφισμα αυτό για το Σύνταγμα και θα κάνει καμπάνια υπέρ του όχι. Αυτό δίνει ε, μια νέα νομιμότητα στην όλη αυτή τη δικασία. Στο οικονομικό μέτωπο η Αίγυπτος αποφάσισε να παγώσει προς το παρόν το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ένα μήνα. Αυτή δεν είναι μια οριστική απόφαση και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κύριοι Ευρωβουλευτές, η Υπάρχει εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Κάθη Άστον, καθώς επίσης και ο Περαδίνο Λεόν, ο ειδικό αντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Κάιρο, ε, έχουν συνεχείς επαφές με τους κύριους πολιτικούς ε, πρωταγωνιστές και με τον Υπουργό Εξωτερικών μεταξύ αυτών. Ε, τονίζουμε σε όλα τα μηνύματά μας την ανάγκη για συμφιλίωση και αποκλιμάκωση. Αυτή είναι η προτιμόμενη δράση για μας λόγω της πόλωσης ε, που υπάρχει μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και της ευαισθησίας που υπάρχει και στις δύο πλευρές σχετικά με την ε, εξωτερική επέμβαση. Όπως ξέρετε, την περασμένη Τετάρτη η ύπατη εκπρόσωπος ε, σε μια δημόσια δήλωσή της ε, τόνιζε πόσο σημαντικό είναι η Αίγυπτος να συνεχίσει την ε, μετάβαση της προς τη δημοκρατία και ζήτησε ένα διάλογο με συμμετοχή όλων. Επανέρχομαι στην αρχική μου ερώτηση σχετικά με τη δημοκρατική μετάβαση της Αιγύπτου. Η οικοδόμηση της ε, δημοκρατίας δεν είναι κάτι που γίνεται στα γρήγορα. Πολλοί από εσά έχετε βιώσει παρόμοια διαδικασία πρόσφατα στις χώρες σας. Ξέρετε ότι η οικοδόμηση μιας βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί σκληρή δουλειά, δέσμευση, ορμή καθώς επίσης και υπομονή. Ε, στο εσωτερικό και στο διεθνές επίπεδο. Μερικές φορές οι δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται, ε, αν τα δει κανείς εκ των υστέρων, ε, δεν ε, είναι σωστά. Όπως είπε κάποιος από τους συναδέλφους τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, η μετάβαση είναι πάντα κάτι το μπερδεμένο και μερικές φορές σημαίνει ότι λαμβάνονται διχαστικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό όμως να λαμβάνονται υπόψη τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι η δήλωση αυτή συνοψίζει την κατάσταση στην Αιγυπτό πολύ καλά. Και τώρα πλέον είναι θέμα της ηγεσία μαζί με την αντιπολίτευση να εμπλακούν σε ένα πραγματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για να βρουν μια συναντητική λύση που θα ανήκει σε όλους ούτως ώστε να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη όσον αφορά τη δέσμευση της Αιγύπτου στην δημοκρατική μετάβαση. Και επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι πρωταρχική σημασίας η Αίγυπτος να αποκτήσει ένα σύνταγμα το οποίο να εκπροσωπεί και να εκφράζει όλους τους Αιγυπτίους που θα εξασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους ανεξάρτητα από την πίστη, το φύλλο ή οποιοδήποτε άλλη παράμετρο. Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πλατεία Ταχύρ και σε άλλα σημεία και ε, ζητώντας και διεκδικώντας τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Κύριοι Ευρωβουλευτές, η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη ε, κατάσταση. Αλλά πρέπει μόνοι τους να βρουν τη λύση. Η Αίγυπτος ανήκει στους Αιγύπτιους. Και εμείς θα δεν θα ε, έπρεπε και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μια λύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το λαό της Αιγύπτου μέσα σε αυτή την δημοκρατική μετάβαση και θα πρέπει να συνεχίσουμε την έκκλησή μας για έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και για μια λύση που θα βασίζεται στη συνένεση. Και ε, απαγορεύοντας βεβαίως οποιαδήποτε μορφή βίας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εκφράσει σαφώς ε, τις προσδοκίες της για μια δημοκρατική μετάβαση και θα, υπενθυμίζοντας ε, την επιτυχή συνάντηση της Task Force με την Αίγυπτο στις 13 και 14 Νοεμβρίου, όπου κάποιοι από εσά ε, συμμετείχατε. Ε, και που είναι η νέα βάση για τις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο με βάση τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Περνάμε στου αγορητέ που θα παρέμβουν εξ ονόματο των κοινοβουλευτικών ομάδων του. Πρώτα απ' όλα θα παρέμβει εξ του ΕΛΚΑ ο κύριος Κριστιαν Πρέντα. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ κύριε Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, Επίτροπε. Θέλω να καλωσορίσω το ότι διεξάγεται η συζήτηση για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Είναι κατεπίγοντος χαρακτήρα αυτή η συζήτηση, διότι αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους ε, η Αίγυπτος. Ε, τα γεγονότα ε, εκτιλήσονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε προς τον εκδημοκρατισμό, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δυστυχώς, με κάθε μέρα που περνά, εκφράζω τη θλίψη μου γι' αυτό, απέχουμε όλο και περισσότερο από αυτόν τον ευκταίο στόχο και βλέπουμε και το διάταγμα, πρόσφατο διάταγμα που είναι απόδειξη αυτών των γεγονότων. Επιτρέπεται οι ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός της Αιγύπτου να συλλαμβάνει πολίτες και να τους προσαγάγει σε στρατοδικεία για να δικαστούν. Ενώ είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Μόρση απέσυρε το διάταγμα το οποίο θα του έδινε υπερεξουσίες μετά όμως από δύο εβδομάδες δισταγμών και πιέσεων που ασκήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν ήταν τόσο κατακαιρματισμένοι και διχασμένοι οι πολίτες της ε, Αιγύπτου όπως σήμερα. Δεν είναι μόνο τα θέματα του ίδιου του Προέδρου Μούρση που τους διχάζουν. Υπάρχει μεγαλύτερος διχασμός και για τον ρόλο της θρησκείας στη δημόσια ζωή, στο δημόσιο βίο και πώς θα είναι δυνατόν να έχει γεφυροποιηθεί αυτό το χάσμα με την επιβολή ενός συντάγματος με αυτές τις διαργασίες. Ιδιαίτερα αν συνταχθεί αυτό το σύνταγμα χωρίς ευρύτερο πλαίσιο διαβουλεύσεων και συζητήσεων και ιδιαίτερα όταν δεν θα υπάρχει κανένα ηχέγγυο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή να πάψουν αυτές οι αυταρχικές δεσποτικές τάσεις από πλευράς ε, των ε, Αιγυπτιακών αρχών. Η μόνη αντιμετώπιση της κρίσης, η μόνη διέξοδος είναι το να συμπεριλάβουν περισσότερους πολίτες στην πολιτική διεργασία για να υπάρχει δημοκρατικός χαρακτήρας και για την ακύρωση των διαπραγματεύσεων ε, βραχυπρόθεσμα ξαφνικά από τις στρατιωτικές αρχές με τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους και παρόλα αυτά θα συνεχίσουν συνεχιστούν οι διεργασίες και θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα παρόλο το κλίμα σύγχυσης που επικρατεί και αυτή τη σύγχυση που έχει επιβληθεί ακόμα σύγχυση και για την ίδια την ημερομηνία κατά την οποία θα γινόταν αυτό. Και δυστυχώς επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Αίγυπτο είναι πραγματικά ένα, μια φάρσα, μια δημοκρατική φάρσα και καθόλου δημοκρατική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Στη συνέχεια ο κύριος Παντσέρη, εξ ονόματος των σοσιαλιστών συναδέλφων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πολιτική φάση αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο είναι κάτι που θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του συναγής. Για αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες πρέπει να εκφράσουμε την αξιολόγησή μας και να καθορίσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές εκτός από την ε, χρονολογική ε, απαρίθμηση των γεγονότων. Ε, από την έκβαση της κατάστασης στην Αίγυπτο εξαρτάται η ισορροπία ολόκληρης της περιοχής, ιδίως και μετά τη δύσκολη αγεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά οι δράσεις ε, του ε, Αιγύπτιου Προέδρου δημιούργησαν πολλά δημοκρατικά προβλήματα και προκάλεσαν τη δίκαιη αντίδραση τη αντιπολίτευση. Πρέπει να είμαστε σαφεί, χωρί να επέμβουμε, αλλά να είμαστε σαφεί. Δεν είναι δυνατόν να φανταστεί κανεί ότι η δημοκρατική μετάβαση τη Αιγύπτου θα γίνει μέσα από τέτοιε χειραγωγήσει, ε, κυρίω ε, μέσω τη λογική ότι όποιο έχει την πλειοψηφία έχει απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει για τη συνταγματική πορεία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν μπορούμε να να μην πούμε ότι το κείμενο του συντάγματος έχει πάρα πολλές ελλείψεις, είναι συντηρητικό και δεν εκφράζει ολόκληρη την κοινωνία της Αιγύπτου. Πρέπει να εργαστούμε ε, ώστε να ξαναρχίσει ο διάλογος και για να γίνει μια σωστή διαχείριση της ε, μεταβατικής φάσης με ουδέτερο ρόλο ε, των ένοπλων δυνάμεων. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να ε, γυρίσει προς τα πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια πολύ πιο ισχυρή παρουσία γιατί πριν και από τις ΗΠΑ η Ευρώπη έχει κάθε συμφέρον να ολοκληρώσει ειρηνικά η Αίγυπτος τη μετάβασή της προς τη δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά η κυρία Σάκε, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε, αυτή είναι μια έκκληση ε, για από την κυρία Άστον. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε ε, στους πολίτες μας και στην Βόρεια Αφρική που ήθελαν δικαιοσύνη, ελευθερία. Είδαμε τις συνέπειες που υπο, της υποστήριξης δικτατορικών καθεστώτων με αβέβαιο μέλλον. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πολιτική που να βασίζεται σε αξίες ε, για συμφωνίες ε, και να υπάρχουν ε, δεν εφαρμόστηκε η πολιτική για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τώρα δοκιμάζεται η πολιτική αυτή. Ο κύριος Μόρση έκανε πολύ κακή κρίση ε, και ήθελε περισσότερη εξουσία από ό,τι είχε ο πρόεδρος Μουτμπάρακ. ήθελε να τεθεί εκτός του δικαστικού ελέγχου οι προσπάθειες ε, οικοδόμησης οικονομικής αντικαταστάθηκαν με κατεπίγουσες πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης. Ο λαός της Αιγύπτου δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Η δημοκρατία είναι κάτι ε, περισσότερο από έναν άνθρωπο που να κυβερνάει. Χρειάζεται κράτος δικαίου. Και ποια ήταν η αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτήν ε, την προδραστική προσπάθεια. Είχαμε μια δήλωση ασθενή και η πρώτη δήλωση μετά τον 22 Νοεμβρίου από την κυρία Άστον ήταν ότι ε, έπρεπε να επιστραφούν στην Αίγυπτο οι παγωμένες κατοθέσεις ε, του καθεστώτος Μουμπάρακ. Ε, δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Η εταιρική σχέση με τη Νέα Αίγυπτο είναι πολύ σημαντική για μας. Ε, όταν οι άνθρωποι ευημερούν στην γειτονιά μας ευημερούμε και εμείς αλλά πρέπει να ζητήσουμε τις οικουμενικές αξίες για όλο το λαό της Αιγύπτου. Είναι απογοητευτικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισχυρότερη ε, διότι είναι σαν να ε, αμελούμε τον λαό της Αιγύπτου. Πρέπει να, είμαστε, να επαγρυπνούμε περισσότεροι ή να πάψουμε να μιλούμε για αιρεσιμότητα. Σας ευχαριστούμε κυρία Σάκε. Εξ ονόματος των Πρασίνων, στη συνέχεια για 1,5 λεπτό, η κυρία Judith Σαρτζεντίνη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όταν ένας φίλος κάνει κάτι περίεργο και κάποιος δεν καταλαβαίνει γιατί το κάνει, τι κάνουμε. Τι κάνουμε όταν προσπαθεί μια χώρα να εκδημοκρατιστεί αλλά πολλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι πλέον εφικτή η υιοθέτηση κάποιων συμβιβασμών. Πρόσφατα είχαμε πάει στην Αίγυπτο με την Task Force ε, και είχαμε συζητήσεις και επιτόπου από πρώτο χέρι και διαπίστωσα ότι ένας συμβιβασμός ε, θα ήταν μια, ένα βήμα προς τα εμπρός ε, έναντι μιας οπισθοδρόμησης ακόμα και αν κάποιος ε, δεν συμφωνεί. Για παράδειγμα, σε σχέση με την αντιμετώπιση ε, του ενός ε, με τον άλλον. Ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ βλέποντας ε, ποιες, θέσεις υιοθετεί ο πρόεδρος Μόρση. Αλλά ακόμα και αν κάνει κάποιος φίλος κάτι το παράλογο, έχει κάποιος το καθήκον ως φίλος να του πει την αλήθεια, ειλικρινά και ξεκάθαρα. Και αν θέλει να περάσει ένα σύνταγμα δια της βίας ο Μόρση, είναι ασύνετο αυτό. Να του το πούμε ξεκάθαρα. Αλλά ταυτόχρονα παραμένουν με φίλοι και παραμένει κανείς φίλος με ένα τέτοιο άτομο και προσπαθεί να υποστηρίξει το φίλο του και να τον συνετίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να μεριμνήσει να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην Αίγυπτο. Όμως μπορεί να βοηθήσει, να συνδράμει τους Αιγύπτιους. Γι' αυτό το μήνυμά μας είναι προς όλους ότι πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε τα πράγματα εκ του Η δημοκρατία όμως όμως δεν μπορεί να αποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Για τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ε, ο κύριος Δόκτωρ Τάνοκ. Γνωρίζουμε ότι μία επανάσταση δεν είναι μία μεταμόρφωση απλή αλλά μία μεταβατική περίοδος ε, και βλέπουμε ότι οι πράξεις του κυρίου Μόση πρέπει να καταδικαστούν. Η σύνταξη του καινούριου συντάγματος θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο εύρος και φάσμα από ότι τις θέσεις και τοποθετήσεις ε, των μουσουλμάνων αδερφών. Ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι προσπάθησε να επεκτείνει με καταχρηστικό τρόπο τις εξουσίες του ο πρόεδρος Μόρση και να ε, υποβάλει, να επιβάλλει τις απόψεις του και στους δικαστές. Και υπάρχει αντίσταση και αυτό το οποίο συνέβη τώρα είναι μια μερική ανατροπή αυτού του προηγουμένου διατάγματος. Ακούσαμε ότι η αντιπολίτευση θα συμμετάσχει λέει στο μελλοντικό δημοψήφισμα και δεν θα το μποϊκοτάρει. Και χαιρετίζεται η ομάδα εργασίας της ε, Λέδισα Άστον που υπόσχεται να συνδράμει τους Αιγύπτιους στον εκδημοκρατισμό. Και σέβονται, ε, λένε ότι θα σέβονται τις ε, θρησκευτικές ελευθερίες των κοπτών και έναντι των απειλών των μουσουλμάνων αδερφών και της Σαρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε και εξ ονόματος ε, της Ευρώπης για τις Ελευθερίες και τη Δημοκρατία ένα λεπτό κύριο Μπάστιαν Μπέλντερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε από τις συζητήσεις που κατά το τελευταίο διάστημα και αυτή την εβδομάδα είχαμε την χριστιανική μειονότητα στην Αίγυπτο με σαφή τρόπο μπορώ να συναγάγω το συμπέρασμα ότι οι χριστιανοί θεωρούν αυτό το νέο σχέδιο συντάγματος κάτι το οποίο πρέπει να απορριφθεί κάθετα και δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη θέση μια προσεκτική ανάγνωση του κειμένου του συντάγματος αποσαφηνίζει γιατί και οι χριστιανοί αλλά και οι υπέρμαχοι ενός κοσμικού λαϊκού κράτους είναι κατά αυτού του σχεδίου συντάγματος. Ένα παράδειγμα, ένα άρθρο αυτού του συντάγματος ε, καθιστά την κωδικοποίηση και την εφαρμογή σε πλήρης διαστάσεις της Σαρία, του θρησκευτικού δηλαδή νόμου του Κορανίου. Και στο άρθρο 4 εκεί συνιστάται στο ανώτατο συμβούλιο να είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της συνταγματικότητας αυτών των διατάξεων και για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται ο θρησκευτικός νόμος, η Σαρία. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα και αυτά υπαρκούν. Ποια συμπεράσματα θα συναγάγουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο από αυτό το σχέδιο, αυτό το εγχείρημα του κυρίου Μόρση που είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή της Αιγύπτου, που είναι ο μόνο, μόνο ηγέτης της μουσουλμανικής αδερφότητας. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια για την Ενωτική Αριστερά, η κυρία Μαρίζα Ματίας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Μόρση και οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν ε, ιδιοποιηθεί του, ε, της άνοιξης, της αραβικής άνοιξης και έχουν επιβάλει ένα δεσποτικό καθεστώς και σε σχέση με την προσφυγή στις ένοπλες δυνάμεις ε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είναι μηνύματα μιας πολύ ανησυχητικής εξέλιξης. Ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος Μόρση και οι αδερφοί μουσουλμάνοι προσπαθούν να καταστήλουν τις ε, διαδηλώσεις δείχνουν την, τον αυταρχικό χαρακτήρα του καθεστώτος με την υποστήριξη των στρατιωτικών. Και πάλι εδώ οι στρατιωτικές δυνάμεις εμπλέκονται στην καταστολή. Το να χρησιμοποιεί κανείς τις στρατιωτικές, τις ένοπλες δυνάμεις για να καταστήλει τις ε, διαδηλώσεις είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο που κάνει η κυβέρνηση Μόρση αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπήρξε μια οπισθοδρόμηση όσον αφορά την θέση των δικαστών. Όμως η προσπάθεια ταχύτατα να επιβληθεί ένα σύνταγμα μέσα σε 19 ημέρες δείχνει ότι είναι πολιτικά πολύ ικτρή η κατάσταση αυτής της χώρας. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με τις πρώτες εκλογές που είχαμε δύο υπαλλήλου, δύο υποψηφίους και τώρα ε, θα έχουμε ε, ακόμα μικρότερη ε, συμμετοχή. Αυτό θα δικαιολογούσε πραγματικά εξέταση των συνταγματικών θεμάτων και εμβάθυνση σε αυτά. Δεν έγινε αυτό. Ελπίζουμε να μην επανέλθει η Αίγυπτος και οπισθοδρομήσει σε τέτοιες σειράξεις. Και πραγματικά πρέπει να δώσουμε την υποστήριξή μας στους Αιγύπτιους. Ευχαριστούμε Μαρίζα. Ολοκληρώνουμε αυτό το γύρο με την παρέμβαση του κυρίου Μέλτσερ. Ένα λεπτό έχει ο κύριος Μέλτσερ για να μας μιλήσει εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Μόρση το ότι ε, υπάρχει ένα επίμαχο σύνταγμα στο οποίο υπάρχουν πολλές ε, αντιδράσεις ε, μπορεί να το εκλάβει κανείς ένα πρώτο βήμα προς μια Ισλαμική δικτατορία απέτυχε αυτή η ανατροπή αυτή η επανάσταση δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία για το ρόλο της θρησκείας ε, στη χώρα είναι σαφές ότι αυτή η αραβική επανάσταση είναι ένα πραγματικά ε, πολύ επικίνδυνο ε, παιχνίδι που παίζεται, ένα βαρέλι με πυρίτιδα, με μπαρούτι που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εκραγεί. Και εδώ υπάρχουν οι ανησυχίες των ανθρώπων. Αυξάνεται διαρκώς η ανεργία και τίποτα δεν γίνεται για να αντιμετωπιστεί. Για να αποφευθεί ένας ε, εμφύλιος πόλεμος δεν επαρκεί να χαρακτηρίζει κανείς εχθρούς τους αντιπάλους. Και η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης μελλοντικά πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ανθρώπων των χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. πρόεδρο. σας ευχαριστώ κύριε Μέρτσερ και περνάμε τώρα στον γύρο των παρεμβάσεων που ολοκληρώσαμε τώρα τον γύρο των παρεμβάσεων εξ ονόματος των ομάδων, τώρα θα παρέμβουν οι συνάδελφοι ατομικά. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μαρία Γκαμπριέλη. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ για την παρέμβασή σας κυρία Γκαμπριέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί και με περισσότερο θάρρος να υιοθετήσει θέσεις σαφείς στο ύψος των αξιών μας. Επαγρύπνηση και διάλογος, δύο λέξεις κλειδιά. Είναι σημαντικό να απευθύνουμε μηνύματα Πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα στην κυβέρνηση της Αιγύπτου. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο δεσμευτήκατε για την δημοκρατία. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Νέο σύνταγμα, εκλογές, ε, καλή θεσμοί. Βρισκόσαστε στον καλό δρόμο. Να μην ε, υποκύψετε στα παλιά κλαστικά, τα αυταρχικά, διότι οι πολίτες ε, σας έχουν εμπιστοσύνη. Δεν μπορείτε να τους παρεβλέψετε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να συνοδεύσουμε την Αίγυπτο με τον πολιτικό διάλογο. Δεν είμαστε εδώ για να κατακρίνουμε την κυβέρνηση της Αιγύπτου, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Στο λαό ένα μήνυμα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία των πολιτών που θέλουν να ζήσουν σε μια δημοκρατία που προασπίζεται τα συμφέροντά τους και εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους όλοι οι διεθνείς πρωταγωνιστές θα πρέπει να προωθήσουν ένα κράτος που να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και που θέλει να προοδεύσει. Με την συμπερίληψη των γυναικών στην διαπραγμάτευση και σε θέσεις υψηλού επίπεδου. Ας μην ξεχνούμε τους νέους. Χάρη στο δυναμισμό τους και στην πρωτοβουλία τους μπορεί να κερδίσει η Αίγυπτος επενδύοντας τους νέους. Και ένα μήνυμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ο βασικός εμπορικός εταίρος και η πρώτη πηγή βοήθειας και επενδύσεων. Πρέπει να παίξουμε έναν πρωταρχικό ρόλο. Η Task Force ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αίγυπτο με πρώτη συνεδρία στις 14 Νοεμβρίου στο Κάιρο είναι μια απτή απόδειξη ενισχυμένης συνεργασίας. Και να... Αν μπορείς να μ' ακούσεις Μαρία, μπορείς να μ' ακούσεις. οι διερμηνείς μου λένε ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ταχύτητά σου, αν μπορείς λίγο να επιβραδύνεις συγγνώμη στους Γερμινείς και τους ευχαριστώ. Θα συνεχίσω. Η Task Force ανάμεσα στην Ένωση και στην Αίγυπτο με πρώτη συνάντηση στις 14 Νοεμβρίου στο Κάιρο είναι απτή απόδειξη της ενισχυμένης συνεργασίας μας και αποτελεί επίσης ένα μοναδικό μέσο για επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η προαγωγή της ειρήνης, σταθερότητας και της ευημερίας όπως και των θεμελιωδών αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Αυτή η Task Force θα πρέπει πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους τους παίκτες της δημοκρατικής μετάβασης και να προσδιορίσει ποιοι θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου στην οικονομία και την πολιτική. Έτσι μπορούμε να αγκιστρώσουμε ε, την δημοκρατία και να μην την ξεχνούμε στην ανόρθωση της οικονομίας, στην απασχόληση και στις επενδύσεις συμφέρουσες για όλους. Η εταιρική μας σχέση ενισχυμένη με την Αίγυπτο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά είναι σημαντικό ο διάλογος και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι το στοιχείο κλειδί στην διαδικασία μετάβασης της Αιγύπτου. Σε ευχαριστούμε Μαρία. Τώρα για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο η κυρία Αναγκόμες παρακαλώ. Η Αίγυπτος βρίσκεται μπροστά σε μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση αυτή τη στιγμή μπροστά σε ε, μια μεταβατική ε, περίοδο εκδημοκρατισμού. Οι ένοπλες δυνάμεις ε, αναλαμβάνουν ρόλο που είναι ασύμβατος με τον εκδημοκρατισμό. Ο πρόεδρος έκανε λάθος ο πρόεδρος Μόρση και θα έπρεπε να υπάρχει διάλογος με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που αναφύονται. Ιδιαίτερα με εκείνους που διαδηλώνουν στην πλατεία Ταχρήρ εναντίον ενός σχεδίου συντάγματος που δεν δίνει καμία εγγύηση για ένα κράτο δικαίου, για μια δημοκρατία, ένα δημοκρατικό καθεστώ και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή είναι δυνατόν η πλειοψηφία των πολιτών να αγνοηθεί, οι γυναίκε, οι θρησκευτικέ μειονότητε και σε σχέση με το δημοψήφισμα το οποίο βιαστικά θέλει ο Μόρση να υιοθετηθεί είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Δεν συνεισφέρει να υπάρξει νομιμοποίηση για την κυβέρνηση. Πρέπει να αποφύγουμε την οπισθοδρόμηση σε ένα δεσποτικό Πρέπει να αποφύγουμε τη βήθηση της Αιγύπτου ε, στην ε, ε, θρησκευτική δυσανεξία και στο μίσος. Πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε η τάξη και γνωρίζουμε στην Ευρώπη από τα ίδια τα βιώματά μας και την πείρα μας ότι η μεταβατική εκδημοκρατι... περίοδος εκδημοκρατισμού παίρνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να γίνει εν μια νυχτή. Αυτό απαιτεί να τηρήσει η Αίγυπτος τις υποσχέσεις σχέσεις για τη δημοκρατία και την ελευθερία γιατί υπήρξαν τόσα θύματα για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και θα πρέπει σαφώς να ε, δούμε ότι αυτοί οι οποίοι δίνουν τον αγώνα για τη δημοκρατία στην Αίγυπτο πρέπει να κάνουν το μόρση να σεβαστεί τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των Αιγυπτίων. Δεν ήθελα να στο πω πιο πριν, αναγκόμε, ε, αλλά δεν μπορούσαν να σε παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Θέλω να παρακαλέσω όλου όσου θα παρέμβουν στη συνέχεια να επιβραδύνουν λίγο τι παρεμβάσει του και να μην ε, εκφωνούν τον λόγο του με τέτοια ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται έτσι οι διερμηνεί που είναι πολύ καλοί στη δουλειά του, εξαιρετικοί στη δουλειά του, αλλά δεν μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε δύο λεπτά, να πούν αυτά τα οποία πρέπει να λέγονται σε τέσσερα λεπτά. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη υπόψη και τον πλούτο της επικοινωνίας και τις ανάγκες σωστής επικοινωνίας. 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Ντεσαρνές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε όλοι ότι η κατάσταση είναι σοβαρή στην Αίγυπτο, η οικονομική έχει καταβυθιστεί, έχουμε μια κρίση πολιτική, θεσμική, συνταγματική, δημοκρατική και εγώ πιστεύω ότι οι ερωτήσεις μας και οι αμφιβολίες μας είναι νόμιμες. Θα πρέπει ε, να θέσουμε ερωτήσεις για αυτό το κείμενο το οποίο θα είναι το αντικείμενο του δημοψηφίσματος διότι αφήνει ανοιχτή πόρτα σε όλες τις ερμηνείες και σε όλες τις καταχρήσεις προς την ισότητα ανδρών γυναικών, ως προς την προστασία ε, των ε, μειονοτήτων, των δημοσίων ελευθεριών. Διερωτώμε και διερωτώμε για το κλίμα. Το κλίμα όπου βλέπουμε βία, ε, που βλέπουμε μεγάλους διχασμούς ανάμεσα στους φιλοϊσλαμιστές, ε, σε αυτούς που είναι κατά των Ισλαμιστών. Αυτό το κλίμα δεν είναι πρόσφορο για δημοψήφισμα. Δεν έχουν ενημέρωση οι πολίτες για το δημοψήφισμα. Αυτό μας το έλεγε ένας μπλόγκερ χτες στο τηλέφωνο και 40% των δικαστών δεν θέλουν να επιτηρήσουν αυτό το δημοψήφισμα. Διερωτώμεθα λοιπόν ο πρόεδρος Μόρση θα πρέπει να καθησυχάσει τους πολίτες, να συνεχίσει το διάλογο, την διαβουλεύσεις να ακούσει τις ανησυχίες της νόμιμες της αντιπολίτευσης και να κάνει μια χειρονομία ε, αναβάλλοντας ίσως ε, την ημερομηνία ε, του δημοψηφίσματος. Δεν πρέπει να πράγει τα πράγματα με βία, με εξαναγκασμό και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε κυρία Υπουργέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί τίποτα να επιβάλλει. Ναι, βεβαίως δεν μπορεί τίποτα να επιβάλλει, αλλά μπορεί να μιλήσει και να υπενθυμίσει στεναρά τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό κύριο συνάδελφος Προβέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, οι προθέσεις του Προέδρου Μόρση και των αδερφών μουσουλμάνων είναι πλέον σαφείς. Ένα σχέδιο συντάγματος που δίνει κυρίαρχο ρόλο στη Σαρία σαν πηγή δικαίου και ένα ε, διάγελμα του ίδιου του Προέδρου που το θέτει υπεράνω του νόμου. Ε, ο Μαχμέτ Μπαντέι, ο αρχηγός των αδελφών ε, ε μουσουλμάνων, ε, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, ότι το τζιχάντ είναι ανοιχτό για όλους τους μουσουλμάνους και ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πάρουν τα όπλα εναντίον της Δύσης. Ε, η ε, Αίγυπτος ακολουθεί ένα η κυβέρνηση στην ε, Αίγυπτο ακολουθεί ένα όλο και πιο ολοκληρωτικό δρόμο ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των νέων, των γυναικών κλπ και ο κίνδυνος είναι να αποσταθεροποιηθεί ολόκληρη η περιοχή πρέπει να δώσουμε χωρίς όρους την υποστήριξή μας σε μια δημοκρατική μετάβαση η οποία αποδεικνύει ότι είναι όλο και πιο δύσκολη και γεμάτη από αντιφάσεις. More for more, όπως είπε ο επίτροπο ε, Φίλε. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τι ε, γνήσια δημοκρατικέ ε, δυνάμει που στην Αίγυπτο θέλουν την πραγματική ανανέωση. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό κύριο Βιγγένιν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν παρακολουθώ τι ειδήσει, Έχω μια στην Τεζαβίου ότι όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ε, Διαδηλωτέ στην πλατεία ταχύ, ο στρατό πάλι στου δρόμου. Μέσα σε, δύο, σε λιγότερο από δύο χρόνια έγινε ένα πλήρη κύκλο στην ιστορία. Όμω δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Όλοι πια έχουμε διδαχθεί από την ιστορία. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα και σε στενή συνεργασία ε, με τι ΗΠΑ. Πολιτείες. Ε, στα μέσα του Νοεμβρίου με την επιτυχή Task Force είδαμε ποιε θα ήταν οι σχέσει μα αν ήταν σεβαστή η δημοκρατία και συνεχιζόντουσαν οι δημοκρατικές ε, μεταρρυθμίσει. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή μα όταν απειλείται ε, η δημοκρατία και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις. Είναι μια κρίσιμη στιγμή που ακόμη μια φορά δοκιμάζεται η αξιοπιστία μας. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων απλώς ε, ε, έκανε ένα απολογισμό των εξελίξεων στην Αίγυπτο χωρίς να καταλήγει σε κανένα συμπέρασμα ή σύσταση μια τέτοια στάση δεν μπορεί παρά να ενθαρρύνει αυτούς που έχουν πάρει αυτόν τον ε, ε, επικίνδυνο δρόμο. Ε, σε λίγες μέρες η Αίγυπτος θα αποκτήσει ένα αμφίβολης αξίας σύνταγμα που θα είναι η βάση για όλες τις περαιτέρω εξελίξεις. Απλώς θα λάβει γνώση και πάλι το Συμβούλιο ή θα τοποθετηθεί. Ξέρω πολύ καλά ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να χτίσει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά δεν μπορώ να παραστήσω ότι ε, είμαι τυφλός απέναντι σε εξελίξεις που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Ζιόμπρο, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, τα γεγονότα στην Αίγυπτο δείχνουν ότι η πολιτική ε, της Λέιδης Άστον δεν έχει καμία επιτυχία. Προσκρούει σε δυσκολίες ε, αυτοί που είχαν καταδείξει την απειλή των Ισλαμιστών που θέλαν να καπηλευθούν την δημοκρατική διεργασία στην Αίγυπτο εδώ και ένα χρόνο επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο. Παρακολουθούμε ε, την κατάσταση στην Αίγυπτο και βλέπουμε ότι ο πρόεδρος ε, Μόρση πάει και πέραν των όσων συνέβησαν στο καθεστώς Μουμπάρακα είναι νομίζω κάνει έκκληση λέει Διάστον για τις ε, δυνάμεις ε, που είχαν πάρει την εξουσία ε, στην Αίγυπτο. Έχουμε όμως αρνητικά αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές πρέπει να υπάρξει μια σαφής θέση χωρίς αμφισβήτηση απέναντι στις ενισχυτικά μηνύματα που μας φτάνουν κάθε μέρα από την Αίγυπτο. Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία απειλείται. Ο κύριος Μπόρι Ζάλα για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, η επανάσταση δεν τελείωσε στην Αίγυπτο. ένα σύνταγμα είναι μια μάχη, ένα πεδίο μάχης ε, πεπιθήσεων και αξιών. Ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Αίγυπτο με τις ε, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης που επέστρεφαν στη δημοκρατία. Ε, η Αιγυπτός αντίθετα ποτέ δεν, μπορούσαμε να, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα ε, μοντέλο δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Αν η Αιγυπτός γίνει ένα κράτος χωρίς μυσαλλοδοξίας αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή για τη δημιουργία δημοκρατίας και κράτους δικαίου στο μέλλον. Ελπίζω ότι η Αίγυπτος θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία επιτυχία. Η Ευρώπη χρειάστηκε 200 χρόνια για να επιστρέψει στη δημοκρατία. Παίρνουμε στη διαδικασία Catch the Eye του Προέδρου. Το λόγο. Έχει το λόγο, ε, το λόγο συγγνώμη, έχει η Ελένα Μπασέσκου για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Θεωρήσαμε ότι με την εκλογή του νέου Προέδρου θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Δυστυχώς όμως τις δύο τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Η απόφαση του Προέδρου Μόρση μπορεί να αποτελεί απειλή για το μέλλον της χώρας. Παρακολουθήσαμε όλες τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης, συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου. Γι' αυτό θα πρέπει ο πρόεδρος της Αιγύπτου να μην ε, αποφασίσει υπέρ της επέκτασης των εξουσιών του. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι με το δημοψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου και με το νέο σύνταγμα θα γίνει και ένα νέο βήμα για την μετάβαση προς τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Κατά το catch the eye δεν υπάρχει μπλε κάρτα. Λυπάμαι. Δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία κατά, την, ε, κατά το catch the eye. Ο κύριος Μέρφυ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσοι είχαν ξεγράψει την Αραβική Άνοιξη ε, αποδείχθηκαν λάθος από τις ε, διαδηλώσεις που ακολούθησαν την απόπειρα του Πρόεδρου Μόρση να υπαρπάξει την εξουσία. Βεβαίω, όλα αυτά που κάνει φέρνουν στο νου το Μουμπάρακ, αλλά η απάντηση των νέων και των εργαζομένων δείχνουν πως ε, δεν έχει χαθεί δυνατότητα κινητοποίησης. Η κατάσταση είναι βεβαίως κρίσιμη οι επιθέσεις ε, γυναίκες ε, συνδικαλιστές ε, αυξάνονται και μόνο με μαζική οργάνωση μπορούμε να υπερασπιστούμε όσα έχουν κατακτηθεί και να προωθηθεί η επαναστατική διαδικασία για να τελειώσει η φτώχεια και ο αναλφαβητισμός, για να υπάρχει δωρεάν υγεία και παιδεία για συντάξεις, δουλειές και αξιοπρεπείς μισθούς. Αυτά τα και δικαιώματα δεν θα τα παραχωρήσουν οι καπιταλιστές ε, αδελφοί μουσουλμάνοι, οι φιλελεύθεροι ή ο στρατός. Απλά θα πρέπει να μην υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ιδιωτική περιουσία. Πρέπει να υπάρξει μια, ένας αγώνας για σοσιαλιστική αλλαγή. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Oh, sorry about this. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος φλέγεται. Κυρία Υπουργό, κύριε Επίτροπε, ποιον εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο. Το Μόσρι, τον Αμπρεμούσα, τους αλαφιστές, το στρατό. Ποιον εμπιστευόμαστε. Ιστορικά, αν δούμε την ιστορία της Αιγύπτου, ήταν ο στρατός αυτός ο οποίος στη μεταβατική περίοδο παρενέβη και έβαλε κάποια πράγματα στη σειρά. Τεχνική υποστήριξη αυτή τη στιγμή όποιον κρίνει η παγκόσμια κοινότης ότι μπορεί να επιφέρει την τάξη, τεχνική υποστήριξη χρειάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά και ο κόσμος που βλέπουμε στους δρόμους δεν είναι μόνο ιδεολογικό αυτό, είναι θέμα επιβίωσης η τεχνική μας υποστήριξη εφόσον όπως είπατε κυρία υπουργό η αίγυπτος θα καθορίσει Δεν ξέρω κατά πόσο πρόκειται για μπλε κάρτα ή catch the Να ξέρετε ότι έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κυρία Μουνίθ. Ούτε καν ένα λεπτό χρειάζομαι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διαδικασία του δημοψηφίσματος και το ε, γεγονός ότι η αντιπολίτευση ε, δεν δέχτηκε αυτή τη διαδικασία ε, αποκλεισμού. Επίσης, ε, ορισμένοι διεθνείς παρατηρητές δέχτηκαν να ακούσουν και να παρευρεθούν μάλλον στη διαδικασία του δημοψηφίσματος και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ε, συνοψίσει. Όχι με συγχωρείτε. Από το Συμβούλιο θα ήθελα να ζητήσω να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος πάντα ήταν πάρα πολύ στενή εταίρη που του συνέδε η ιστορία, η γεωγραφία και ο κοινό στόχος ε, σταθερής ε, και ειρηνικής ε, γειτονίας. Εντυπωσιαστήκαμε όλοι όταν Αιγύπτιοι από όλες τις τάξεις βγήκαν στους δρόμους τον Ιανουάριο του 2011 ζητώντας δυνατά και καθαρά τα νόμιμα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε γρήγορα την ομόθυμη στήριξή της σε μια δημοκρατική μετάβαση. Ναι, ο δρόμος ήταν δύσκολος και θα συνεχίσει να είναι δύσκολος πριν οριστικοποιηθεί η δημοκρατική μετάβαση που θα διασφαλίζει ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Όλες είναι Επιχορηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει τώρα να ακολουθούν τις νέες ευρωπαϊκές αρχές όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την Αραβική Άνοιξη. Η νέα αυτή προσέγγιση έχει στόχο να δώσει επιπρόσθετη στήριξη στις χώρες εκείνες οι οποίες πραγματικά εδρεώνουν πολιτικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και προσπαθούν για μια ανάπτυξη με ε, συμπερίληψη και των ασθενεστέρων και κοινωνική δικαιοσύνη. Θα φροντίσουμε αυτές οι αρχές να εφαρμοστούν πλήρως σε όλες τις χώρες της γειτονιάς μας και της Αιγύπτου συμπεριλαμβανομένης. Επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα περισσότερα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν τον Αιγυπτιακό λαό και τα πιο ευάλωτα στρώματά του. Ως παράδειγμα, υιοθετήσαμε φέτος στήριξη σε τομεί κλειδιά, όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η απασχολησιμότητα των νέων και η επαγγελματική κατάρτιση. στήριξη επίσης θα διοχετευτεί στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των ΜΚΟ. Η κατάσταση είναι ρευστή στην Αίγυπτο. Αλλάζει ώρα με την ώρα και συμφωνούμε όλοι πως η Αίγυπτος έχει ζωτική σημασία για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περιοχή. Αναφέρθηκε η περιφερειακή διάσταση και η σημασία της Αιγύπτου όσον αφορά την κατάφαση του πυρός στη Γάζα αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Επίσης συμφωνούμε πως θα πρέπει να έχουμε υπομονή γιατί η μετάβαση βεβαίως χρειάζεται κάποιο χρόνο. Πρέπει να φροντίσουμε ο σεβασμός των μειονοτήτων και ειδικά των θρησκευτικών κοινοτήτων και η οικοδόμηση της συνένεσης είναι βασικά στοιχεία της δημοκρατίας της Αιγύπτου. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι το Σύνταγμα, θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της ε, ευρύτερης εθνικής συνένεσης. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που μεταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ε, Αιγύπτιους εταίρους μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τη στιγμή ακριβώς που μιλάμε συζητούνται νέες προτάσεις διαλόγου. Όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, το θέμα δεν είναι η διπλωματία της Ντουντούκας, αλλά το να είμαστε διακριτικοί δεν σημαίνει πως δεν θα είμαστε σαφείς στα μηνύματά μας. Για να δείξουμε ρεαλιστικά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την δημοκρατική μετάβαση της Ένωσης, Υπάρχει μια ομάδα δράσης η οποία οργανώθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου η οποία ε, διαχειρίζεται όλα τα μέσα στήριξης ε, τουρισμό, επενδύσεις, κινητικότητα και βέβαια στήριξη υπομορφή επιχορηγήσεων και δανείων. Οι πρόσφατες πολιτικές αναταραχές δεν μπορούν να επισκιάσουν την επιτυχία αυτής της ομάδας δράσης. Μέσω της νέας σύμβασης με την Αίγυπτο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μοναδική θέση να βοηθήσει την, Αίγυπτη, Αίγυπτο να τηρήσει κάποιες αρχές και αξίες. Και στην ε, τωρινή κατάσταση βεβαίως χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω πως η δημοκρατική μετάβαση είναι μια μακρά διαδικασία και απαιτεί σκληρή δουλειά, δέσμευση, αντοχή και υπομονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τον Αιγυπτιακό λαό στην δύσκολη αυτή μεταβατική περίοδο με αποφασιστικότητα και επιμονή για να επικρατήσει η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Κοζάκου Μαρκουλή. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι Επίσης ε, ένα θέμα στο οποίο θα κάνει δήλωση η πατή εκπρόσωπος ε, της Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και το θέμα είναι η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους